εκεί εφαρμογή των ε, δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας με ε, εισηγητή τον κύριο Κρόιτσμαν και όπως κάνουμε πλέον συνήθως καταρχήν τώρα, κατά παγία αναρχήν, ε, για κάθε νέο φάκελο που ανοίγουμε ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει μια μελέτη αντικτύπου και επομένως ε, τον στρατηγικό σχεδιασμό που έχει ε, βάλει ως βάση για την πρότασή της και την πρόταση που θα εξετάσουμε. Και μέχρι τώρα αυτό έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο και για μας και για την ποιότητα της εργασίας μας. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε και τώρα Υπενθυμίζω ότι η συνεδρίασή μας είναι δημόσια και μεταδίδεται και μέσω του διαδικτύου και ελπίζω οι, ε, όσοι μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο να μπορούν να δουν και τις διαφάνειες. Υπενθυμίζω επίσης ότι έχουμε και ένα newsletter το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε και ε, στο διαδίκτυο καλύπτει τα θέματα ε, επί των οποίων εργαζόμαστε, έχει και τις ημερήσεις διατάξεις των συνεδριασών μας και για τα παρόντα μέλη αλλά και για όποιον θέλει να μα ζητήσει την ετήσια έκθεσή μας για το 2009. Έχουμε ακόμη μερικές ε, ε, μερικά αντίτυπα σε διάφορες γλώσσες και μπορείτε να το ζητήσετε. Ωραία, καλά σας έκανα την ε, promotion λοιπόν. Τώρα θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, αρχίσει την παρουσίασή της. Ο κύριος Αντώνιος Καστρινάκης. Ελπίζω να μην το χάλασα πολύ το όνομά σας στην έκφορα. Εσείς θα παρουσιάσετε λοιπόν την παρουσίαση, μετά θα λάβει το λόγο ο κύριος Κρόιτσμαν και έχουμε και ε, παρόντες ορισμένους σκιώδης συγητάς όπως την κυρία Σαλντεμόζε, Ρούλε και εγώ προσωπικά. Καλό λοιπόν την ε, Γενική Διεύθυνση Ταξούτ να κάνει την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σημαντική για την προστασία της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και χωρίς επιβολή δεν μπορεί να υπάρξει προστασία. Αυτή είναι η βάση για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό για την τελωνιακή επιβολή της προστασίας των δικαιωμάτων αυτών. Θα σας δώσω πρώτα κάποια πλαίσια πληροφοριών πριν έρθω στην ίδια την πρόταση. σχετικά με εμπορικές ροές που ε, παραβιάζουν τα ε, διανοητικά δικαιώματα, ο ρόλος των ε, τελωνίων είναι σημαντικός, διότι με την παρέμβασή τους έχει τη δυνατότητα ο δικαιούχος να προσφύγει, για παράδειγμα, ενώπιον των δικαστηρίων για θέματα παραβιάσεων των διανοητικών δικαιωμάτων του και αυτή τη στιγμή μπουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα παραποιημένα προϊόντα, είναι πολύ δύσκολο πλέον να αναχαιτιστούν, να εντοπιστούν και να κατασχεθούν. Ενώ εάν κατασχεθούν από ε, τα τελωνία και στα τελωνία, είναι δυνατόν με μία νομόνομική νομική διαδικασία να αντιμετωπιστεί πρόβλημα ολόκληρου φορτίου. Το 2010 η... τα ευρωπαϊκά τελωνία σταμάτησαν 80.000 φορτία με πάνω από ένα εκατομμύρια εμπορεύματα. Ένα εκατομμύριο εμπορεύματα. Πολύ περισσότερε περιπτώσει, πάνω από χίλιε φορέ περισσότερε περιπτώσει, πάνω από χίλιε περιπτώσει μάλλον περισσότερε από το, την προηγούμενη χρονιά. Τα δεδομένα που διαθέτουμε δεν είναι ακόμα πολύ αξιόπιστα. Η γενική πάντως εντύπωση είναι ότι το πρόβλημα ε, αυξάνεται. Η παγκοσμιοποίηση τη παραποίηση και η χρήση του διαδικτύου για παραγγελίες κλπ. είναι και σημαντικές προκλήσεις. Ο πρώτος κανονισμός για την τελωνιακή επιβολή της προστασίας των IPR είναι του 1996. Ε, ε, ε, αναθεωρήθηκε το 2004 διορθώνει δημιουργία το 86 και η τελευταία αναθεώρηση ήταν το 2003. Τώρα προτείνονται ε, βελτιώσεις. Στο σχέδιο δράσεως για τα IPR του 2009, Κομισιόν και Συμβούλιο έχουν περιλάβει ορισμένα στοιχεία που πρόκειται να αναθεωρηθούν. Για παράδειγμα, απλοποιημένες διαδικασίες, η αντιμετώπιση μικρών ε, φορτίων, μικρών αποστολών, η καταστροφή, η αποθήκευση, οι στατιστικές, η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού ε, συστήματος εφαρμογών και η ενδεχόμενη επέκταση της, ε, του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Όλα αυτά από το αντικείμενο ε, διαβούλευσης που διεξήχθη το 2010. Οι παρεμβάσεις των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών έχουν περιληφθεί στην μελέτη αντικτύπου που προσαρτάται στην πρόταση της Επιτροπής. Ταυτόχρονα και εκτός από την, παράλληλα μάλλον με την ε, ε, δημόσια διαβούλευση, Ινδία και Βραζιλία ε, προσέφυγαν για, ονομα... για φάρμακα χωρίς εμπορική ονομασία για κατακρατήσεις προϊόντων, φαρμάκων που έγιναν στην Ολλανδία και εξετάστηκε ο κανονισμός 1383 από Ολλανδικά δικαστήρια. Είναι το λεγόμενο, η λεγόμενη κατασκευή κατά πλάσμα που θεωρήθηκε δηλαδή ότι τα φάρμακα αυτά είχαν παραχθεί στην ίδια, στις ίδιες τις κάτω Κατασχέθηκαν ωστόσο εμπορεύματα και καταστράφηκαν ε, φάρμακα ή και επιστράφηκαν στην Ινδία, χώρα προέλευσης του Ινδία και η Βραζιλία έθεσαν ερωτήματα στα πλαίσια της συμφωνίας TRIPS, διότι θεωρούν ότι υπερβαίνει το συνήθες όριο εφαρμογής και παραβιάζει την ελευθερία ε, transit. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε διαβουλεύσεις με την Βραζιλία και την Ινδία και με την Ινδία κατέληξαν σε συμφωνία, σε ένα γενικό μνημόνιο συμφωνίας δηλαδή για τα δικαιώματα και την εφαρμογή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιλάβει τις αρχές αυτές στην πρότασή της, την οποία έχετε δηλαδή μπροστά σας, και να αντικαταστήσει τον τρέχοντα κανονισμό, καθώς επίσης και στο λεγόμενο soft law, το ατελές δίκαιο δηλαδή, και σε ανταλλαγή η Ινδία συμφώνησε να μην ζητήσει την, ε, την ίδρυση πάνελ στον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου μέχρι ότου εγκριθεί η αναθεωρημένη μορφή της, του Μνημονίου Συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνεται σε αλληλογραφία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ινδικού, ε, εμπορίου, του Ινδικού Υπουργείου Εμπορίου το γεγονός απλώς ότι περνούν τα φάρμακα από ε, ευρωπαϊκή επικράτεια από μόνο του δεν αποτελεί επαρκή λόγο για τις τελωνιακές αρχές σε οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε χώρα μέλος ότι τα φάρμακα αυτά παραβιάζουν τα ε, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν όμως υπάρχει, υπάρχουν στοιχεία που ικανοποιούν τις τελωνικές αρχές ότι υπάρχει πιθανότητα να παραμείνουν τα φάρμακα αυτά στην ευρωπαϊκή αγορά αποτελούν επαρκή λόγο για, τα, για τις ελληνικές αρχές να θεωρήσουν ότι τα εν λόγω φάρμακα παραβιάζουν τις διατάξεις προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κλήθηκε να αποφασίσει επί κατασχέσεων τέτοιων φαρμάκων και ακόμη εκκρεμούν ορισμένες υποθέσεις ενώπιον του ΔΕΚ, αλλά είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί με ποιο τρόπο η, γίνεται η εφαρμογή των κανόνων προστασίας των δικαιωμάτων αυτών. Η πρότασή μας έχει τρεις βασικούς στόχους. Πρώτο, να ενισχύσει την ικανότητα των τελωνίων να, επιβάλλουν την προστασία των ε, δικαιωμάτων Δεύτερο, να ανακόψει την μεγάλη αύξηση μικρών αποστολών μέσω διαδικτύου. Τρίτο, να ξεκαθαρίσει τις νομικές αβεβαιότητες γύρω από τον ρόλο των τελωνίων σε ό,τι αφορά την διακίνηση εμπορευμάτων transit και έτσι να επιληθεί και η διαφορά με την Βραζιλία και την Ινδία χωρίς να προκαταλάβουμε οποιαδήποτε μελλοντικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ορισμούς των ε, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η πρότασή μας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ε, στρατηγικής η οποία απηχείται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενιαία αγορά για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις 24 Μαΐου 2011 καθώς επίσης και της πράξης ενιαίας αγοράς. Εν συμπεράσματι θα ήθελα να πω ότι η πρόταση δείχνει την προτεραιότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2012 και επίσης η πρόταση αναμένεται από τους Ευρωπαίους ε, ενδιαφερομένους και από τις χώρες μέλη με, μεγάλη, με μεγάλο ενδιαφέρον. Αποτελεί προτεραιότητα της Πολωνικής Προεδρίας, η οποία την επόμενη εβδομάδα οργανώνει συνέδριο στην Κρακοβία για την προστασία της διανοητικής ευεκτησίας. Τέλος, η πρόταση είναι ζωτική σημασία και για την επίλυση τη διαφορά μέσα στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπόριου. Ελπίζει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν την πρόταση το δυνατόν συντομότερο μέσα στο 2012. Θα ήθελα παρακαλώ να δώσετε το λόγο τώρα στην ε, συνάδελφό μου. Σε ευχαριστώ. Θα ήθελα με τη σειρά μου να σας παρουσιάσω ε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, το σκεπτικό και τη στρατηγική σκέψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προετοιμασία αυτής ε, της πρότασης και τη μελέτη αντικτύπου. Όπως είπε και ο κ. Καστής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει να αντικατασταθεί ο κανονισμός ενισχύ 1383 το 2003 σε ό,τι αφορά τη δράση των τελωνίων ε, κατά των αγαθών που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να αναλάβουν η κατάλληλη δράση. Σε ε, ό,τι αφορά το περιεχόμενο και πριν αρχίσω θα ήθελα να σας δώσω λίγο το ιστορικό. Τι κάνουν τα τελωνία για την επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, εκτίμηση του κινδύνου για να εντοπίσουν τα ύποπτα φορτία που ενδεχομένω να παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια διεξαγάγουν φυσικούς ελέγχους, συνεργάζονται με τους δικαιούχους, ε, τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και ε, ενημερώνουν για την ενδεχόμενη παραβάση. Επίσης, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι λαμβάνονται υπόψη ε, τα συμφέροντα όλων των ε, ε, θεμητών και νόμιμων εμπόρων και η δράση περιορίζεται στην ταυτοποίηση και στην κατάσχεση των φορτίων. Επίσης ο ρόλος είναι να διευκολύνεται μια απλή καταστροφή των παραποιημένων προϊόντων. Θα ήθελα να σας αναφέρω λίγο και να επιστήσω την προσοχή σας στη δραστηριότητα των τελωνίων. Έχουμε τον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν καταγραφεί ε, και την πρόοδο από το 2000 ως το 2010. Ε, βλέπετε λοιπόν από τη γραφική παράσταση ότι τα τελευταία στοιχεία για το 2010 είναι 80.000 καταγεγραμμένες, καταχωρημένες περιπτώσεις για ένα έτος. Δηλαδή έχουμε σταθερή αύξηση κατά σχέση στα σύνορα από τις τελωνιακές αρχές. Γιατί έχει ε, προκύψει αυτή η αλλαγή. Όπως είπα προηγουμένως, το Συμβούλιο στο ψήφισμά του για την παραποίηση και την πειρατεία κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την κείμενη νομοθεσία. Γι' αυτό αναθεωρήσαμε την ισχύουσα νομοθεσία και ε, κάναμε ε, δημόσια διαβούλευση για μελέτη αντικτύπου. Πολλοί είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή. Μεταξύ αυτών είναι ότι έχει αλλάξει το εμπόριο των παραποιημένων προϊόντων από τον τελευταίο κανονισμό και μετά. Βλέπουμε αύξηση και στον όγκο των προϊόντων, αλλά και ε, μια παγκόσμια πλέον και βιομηχανική διάσταση ε, της παραγωγής ε, και του εμπορίου παραποιημένων προϊόντων. Επίσης, είναι και περισσότερα τα προϊόντα στο παρελθόν, πρόκειται κυρίως για είδη πολυτελείας, αλλά σήμερα κάθε κλάδος βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων είναι ε, θύμα ε, παραποίησης, πειρατείας και βλέπουμε όλο και περισσότερα καθημερινά προϊόντα καθημερινής χρήσης να θίγονται. Επίσης και τα δικαιώματα που παραβιάζονται ως προς το φάσμα τους αυξάνονται. Βλέπουμε και μεθόδους ε, διανομής διαφορετικές από ό,τι στο παρελθόν παραδοσιακά οι κατασχέσεις αφορούσαν φορτία σε λιμάνια και σε αεροδρόμια. Σήμερα βλέπουμε έκρηξη ε, στις ταχυδρομικές αποστολές παραποιημένων ε, προϊόντων και όπως βλέπετε και από τις στατιστικές για το 2010 πάνω από τις μισές περιπτώσεις αφορούσαν ταχυδρομικές αποστολές. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι Έχουμε και πολλές, ε, πολλά αντίτυπα, σας ενδιαφέρουν, ε, της έκθεσης ε, πεπραγμένων του 2010 των τελωνίων. Το περασμένο Ιούλιο εξεδόθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έγγραφο αυτό. Επίσης, η αλλαγή χρειάζεται για να επέλθει κάποια νομική διευκρίνηση στις διαδικασίες, για να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας ε, ταυτόχρονα ε, να μην διακυβεύεται το νόμιμο εμπόριο και να προστατεύονται τα βασικά δικαιώματα. Λοιπόν, για τη μελέτη αντικτύπου η σκότ ποιμότητας, η εφετηρία μας ποια ήταν. Αρχίσαμε με μια εκτεταμένη επισκόπηση και αναθεώρηση της ε, βιβλιογραφία, στην παραποίηση, ε, τι σημαίνουν αυτά από τα προϊόντα για την αγορά. Πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι πολλές ε, οι μελέτες και πολλές εκθέσεις, αλλά λίγα τα στοιχεία που είναι αξιόπιστα. Η μεθοδολογία δεν είναι η ίδια, οι μελέτες δεν είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να έχει κανείς μια πάρα πολύ ξαφή εικόνα ε, των παράνομων εμπορικών δραστηριοτήτων. Μελετήσαμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και μια από τις πιο γνωστές μελέτες είναι του ΟΣΑ, όπως γνωρίζετε, το 2007, η οποία αναθεωρήθηκε το 2009 για την παραποίηση στο διεθνές εμπόριο και τα παρεποιημένα προϊόντα και ο ίδιος ο ΟΣΑ παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να έχει αξιόπιστα στοιχεία. Ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραποίηση και την Πειρατεία των Προϊόντων αντιμετωπίζει το θέμα αυτό και έχει αρχίσει και ε, εργασίες για να βρει μια μεθοδολογία που να εκτιμά το μέγεθος και τον αντίκτυπο όλων αυτών στην πραγματική οικονομία. Παρά τις δυσκολίες των στοιχείων, βλέπουμε τρεις τάσεις. Ε, σας είπα, Αυξάνεται ε, ο όγκος ε, των παραποιημένων προϊόντων και βλέπουμε και ολόκληρες εταιρείες ε, που αφιερώνουν πολλά χρήματα στην καταπολέμηση της παραβίασης των πνευματικών τους δικαιωμάτων. αυξάνονται τα προϊόντα και αυξάνεται και η διανομή πλέον μέσω διαδικτύου που είναι σημαντικό στοιχείο πρόκληση ουσιαστικά για τα τελωνία θα πρέπει να ληφθεί ε, άμεση ε, να ληφθεί μάλλον άμεση δράση και στα ε, σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και περιορισμοί και δυσκολίες στην αναθεώρηση της νομοθεσίας. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μια νομοθεσία που ισχύει ήδη από το 1986 όπως υπόθηκε και το σύστημα που έχει εδραιωθεί, ε, λειτουργεί αρκετά καλά πολλές φορές. Οπότε χρειάζεται περιορισμένες ε, αλλαγές. Ε, άλλες δυσκολίες και περιορισμοί είναι οι διεθνείς μας υποχρεώσεις. Όπως γνωρίζετε, αυτό είναι στοιχεία της συμφωνίας TRIPS από το ΠΟΕ. Ξέρετε ότι είναι η συμφωνία του ΠΟΕ για την πνευματική ιδιοκτησία και επίση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Όπως είπε ο κύριος Καστρισιανάκης, ε, κάναμε πέρυσι ευρύτατη ε, δημόσια διαβούλευση με έξι ερωτήσεις. Τι μπορεί να κάνει ε, κανείς για να προστατεύσει ε, την επιβολή των ε, πνευματικών δικαιωμάτων στα σύνορα χωρίς να εμποδίζει το νόμιμο εμπόριο. Το θέμα είναι σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει τα τελωνία να λαμβάνουν δράση για να προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα. Και εδώ μπαίνει και η προβληματική της διαμετακόμισης του ε, στο εμπόριο. Επίσης, ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και, ποια, και πόσα είναι τα δικαιώματα που καλύπτονται. Είναι αρκετά, χρειάζεται μήπως διεύρυνση ε, ο κανονισμός ή περιορισμός στο πεδίο εφαρμογής του. Για τους δικαιούχους και τους ενδιαφερομένους υπάρχουν κάποιες ε, ε ε, θα πρέπει να διατηρηθούν αυτές. Επίσης ζητήσαμε από τους ενδιαφερμένους να μας πούν τη γνώμη τους για την απλουστευμένη διαδικασία, για τις μικρές ε, παρτίδες ή τα μικρά φορτία και το θέμα ε, του κόστους. 89 απαντήσεις λάβαμε από ευρύτατο φάσμα ενδιαφερομένων μεταφορείς, δικηγόρους, πανεπιστημιακούς, ΜΚΟ, πολίτες, κρατικές αρχές κτλ. Από όλες αυτές λοιπόν τις απαντήσεις και από όλα τα θέματα που ρωτήσαμε, γιατί μας το ζήτησε το Συμβούλιο, τα έχουμε συνοψίσει στις τρία βασικά προβλήματα που χρειάζεται να διορθωθούν. Πρώτο πρόβλημα. Ορισμένα πνευματικά δικαιώματα δεν επιβάλλονται από τις τελωνιακές αρχές στα τελωνία. Ας πούμε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με εμπορικά σήματα, ε, με ημιαγωγούς ή και κάποια άλλα στοιχεία που αποκλείονται. Ας πούμε το ε, αθέμητο παράλληλο εμπόριο είναι κάτι το οποίο διαφεύγει σήμερα των τελωνίων. Ε, έχουμε και διάφορα δικαιώματα που παραβιάζονται Όπως μας είπαν οι ενδιαφερόμενοι εταιρείε, ας πούμε, μας λένε ότι πληρώνουν πάρα πολύ ε, μεγάλο τίμημα για να επιβάλλουν τα πνευματικά τους δικαιώματα όταν κυκλοφορεί το προϊόν τους στην ενιαία αγορά. Και θα ήταν πιο φτηνό πριν την κυκλοφορία στην αγορά να δρουν τα τελωνία. Έχουμε λοιπόν τρεις πλέον δυνατότητες και προτάσεις για λύσεις. Η πρώτη πρόταση είναι να μην κάνουμε τίποτα, να παραμείνει η κατάσταση αμετάβλητη και παρόλο αυτό θα έχουμε υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις και το επίπεδο επιβολής στην Ένωση δεν θα βελτιωθεί. Άλλη δυνατότητα είναι τα μη νομοθετικά μέτρα αλλά εμεί δεν μπορούμε να αλλάξουμε το πεδίο του κανονισμού με μη νομοθετικά μέτρα. Και η τρίτη επιλογή ήταν να κάνουμε μια πρόταση για νομοθετική αλλαγή, για νομοθετικά μέτρα να προσαρμοστεί ε, το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού με τον εξή τρόπο. Να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής σε όλα τα πνευματικά δικαιώματα που ήδη καλύπτονται από τον κανονισμό. Παράδειγμα, κάποια εμπορικά σήματα που οδηγούν σε σύγχυση για την αντιγραφέση και το παράλληλο εμπόριο. Και ε, ήδη αυτό από μόνο του ε, είναι αποτρεπτικός παράγον ε, για τις εταιρείε να κυκλοφορούν στην αγορά παραποιημένα προϊόντα τους. Το κόστος όμως για τη διοίκηση και για τους εμπόρους είναι δύσκολο να εκτιμηθεί γιατί αυτές τις προφορίες είτε δεν τις έχουμε σήμερα είτε είναι εμπιστευτικές. Η δεύτερη δυνατότητα είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή σε κάθε είδους παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων που καλύπτει ο κανονισμός, συν όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται μέσα στην Ένωση, αλλά δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Όταν είδαμε όλα αυτά τα επιπλέον δικαιώματα και τα μελετήσαμε, καταλήξαμε ότι δεν θα οδηγήσει σε ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και της επέμβασης των τελωνίων. Το 90% σήμερα ε, γίνεται με ε, τον κλασικό τρόπο. Αν επεκταθεί όμως ο κανονισμός σε όλα αυτά τα δικαιώματα θα μπορούν οι δικαιούχοι να επικαλούνται και να έχουν καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων τους. Ε, ε, αντί να είναι υποχρεωμένα τα τελωνία να αφήνουν τα εμπορεύματα να περνούν γιατί δεν έχουν την αρμοδιότητα να τα σταματήσουν. Θέλουμε λοιπόν καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ένωση και οι ενδιαφερόμενοι και οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να κυνηγούν τα προϊόντα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα διάφορα καταστήματα αλλά να σταματούν αυτά ε, στα σύνορα όταν εντοπίζετε το φορτίο πριν κυκλοφορήσει στην Ένωση. Οι διοικητικέ επίση διαδικασίες που έχουμε σήμερα ε, στην νομοθεσία είναι πολύ βαριέ. και για τους ε, δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και για τα τελωνία. Κοιτάξαμε δύο ειδικά θέματα. Το ένα είναι η απλούστευμένη, απλοποιημένη διαδικασία για την καταστροφή των προϊόντων αυτών. Σήμερα είναι θελοντική αυτή στον κανονισμό που σημαίνει ότι δεν την εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει καταστροφή των προϊόντων χωρίς καμία νομική διαδικασία, χωρίς να έχει προσφύγει λοιπόν ε, στα δικαστήρια ο ενδιαφερόμενος και ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η διαδικασία λέγεται απλοποιημένη θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο και απαραίτητο να ε, εξασφαλιστεί η δυνατότητα αυτή σε όλα τα κρατημέρια, αλλά να γίνει δεσμευτικό αυτό για να εφαρμόζεται. Το άλλο θέμα που μας απασχόλησε ήταν οι πωλήσει ε, των ε, προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Πέρυσι είχαμε 550.000 συγγνώμη, ε, τέτοιες ε, περιπτώσεις. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η διοικητική διαδικασία εξέταση αυτών των προϊόντων, γιατί πολλές φορές είναι πολύ μικρές οι παρτίδες, δεν είναι φορτία, είναι ένα ή δύο προϊόντα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα να μην κάνουμε τίποτα, να αφήσουμε την κατάσταση ως έχει, ε, πράγμα που θα επιδεινωθεί τις μικρές αποστολές και τελικά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον όγκο τα τελωνία και δεν θα προστατεύονται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση διανοητικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ή δίνουμε συγκριτικό πλεονέκτημα σε εταιρείε που εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν μπορούμε να τις ε, διώξουμε και μπορούν να στέλνουν στην ευρωπαϊκή αγορά ε, προϊόντα από το εξωτερικό. Ενώ εταιρείε που έχουν την έδρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχονται αυστηρά. Αν δεν κάνουμε τίποτα, το κόστος της ε, κράτησης ε, θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Και αυτό αφορά και την ε, διαδικασία και τη διαδικασία η οποία έχει μεγάλη διάρκεια. Είχαμε λοιπόν την επιλογή του να μην κάνουμε τίποτα. Υπάρχει όμως και η πρόταση υποβολής νομοθετικών μέτρων έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να γίνει δεσμευτική στα κράτη-μέλη, δηλαδή της υποχρεωτικής καταστροφής έτσι ώστε να γίνει, μια, να γίνει εναρμόνιση στα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μειώσει και τον διοικητικό φόρτο της ε, παρακράτησης της κατακράτησης. In order to the administrative burden for... Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι να δούμε ότι σε, στις ε, περιπτώσεις που υπάρχει παραχάριξη τα τελωνία αποστέλουν μία επιστολή στον ιδιοκτήτη των αγαθών και τον ερωτούν κατά πόσο μπορεί, ε, ε, επιθυμεί μάλλον να αποστείλει το προϊόν για καταστροφή χωρίς να υποστεί κυρώσεις με βάση αυτή τη διαδικασία. Αυτό θα γίνει χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις στον καταναλωτή και χωρίς να επιβαρύνεται ο καταναλωτής, διότι πολλές φορές ο καταναλωτής δρά καλή την πίστη και υφίσταται τις επιπτώσεις. Τώρα, ως προς τα μη νομοθετικά μέτρα θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά δεν μειώνουν το διοικητικό κόστος αυτής της ε, μακροχρόνιας διαδικασίας. Υπάρχει και ένα τρίτο πρόβλημα που είναι το εξής το ότι ορισμένες ε, πτυχές των διοικητικών διαδικασιών θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ώστε να οδηγήσουν σε ε, μία ανισόρροπη προσέγγιση σε σχέση με τους διάφορους, ε, τη θέση των διάφορων εμπλεκομένων φορέων. Και ένα από τα πρώτα ζητήματα τα οποία μας απασχόλησαν έγκυται στο ότι οι διαδικασίες μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της διαμετακίνησης των φαρμακευτικών ε, σκευασμάτων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπάρχει η δυνατότητα του να μην κάνουμε τίποτα και στη συνέχεια θα μπορούσαμε να ε, ακολουθήσουμε την πολιτική αντιμετώπισης του θέματος με βάση την οδηγία των περιφαρμακευτικών σκευασμάτων. Ως προς την ε, νομοθετική προσέγγιση θεωρούμε ότι ε, δεν θα μας οδηγήσει στο τέλος της διένεξης στα πλαίσια του ΠΟΕ. Επίσης μιλάμε για νομοθετικά μέτρα για να διορθώσουμε την κατάσταση ασαφιών Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ε, μεγάλη διαφορά ή αν υπάρχει διαφορά μπορεί να επιληφθεί σε επίπεδο ΠΟΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Επίσης, το δικαίωμα της υπεράσπισης δεν έχει εγγραφεί σε αυτόν τον κανονισμό, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να ενταχθεί στην περίπτωση των τελωνίων που ε, παρακρατούν τα αγαθά έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορέσει να προβάλλει την υπεράσπισή του. Επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα της απλουστευμένης καταστροφής όταν τα τελωνία αποφασίσουν για τη στραφή καταστροφή των αγαθών με βάση την απλουστευμένη διαδικασία θα πρέπει να ζητήσουν από τους εμπλεκόμενους φορείς να συμφωνήσουν για αυτή την καταστροφή. Και εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε να μην κάνουμε τίποτα, οπότε θα υπάρχει ασάφεια δικαίου, είτε να προβάλλουμε νομοθετικά μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση. Αυτά ως προς την μελέτη επιπτώσεων. Στη συνέχεια το υπόλοιπο της παρουσίασης αφορά την πρόταση αυτή. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα να δείτε εσείς τις διαφάνειες που αναφέρονται σε όλα τα ζητήματα και που αναγράφονται στην πρόταση της Επιτροπής Και μετά για να κατανοήσετε καλύτερα την πρόταση έχουμε μία περιγραφή, την περιγραφή των διαφόρων κεφαλαίων και νομίζω ότι θα έχουμε και άλλη, μία, άλλη δυνατότητα, μία μελλοντική δυνατότητα να επεκταθούμε στα επιμέρους θέματα που αποτελούν την μελέτη αντικτύπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί μας σκιαγραφίσατε ορισμένα βασικά ζητήματα που αφορούν αυτό το τομέα. Μας δώσατε και το ιστορικό, το οποίο βοηθά ιδιαίτερα και ίσως θα ήταν σκόπιμο να ασχοληθούμε και με θέματα παραπομπής στον ΠΟΕ γιατί υπάρχουν ορισμένα ευαίσθητα ζητήματα τα οποία δυστυχώς πρέπει να παραπεμφθούν εκεί. Δεν επιλύονται εύκολα οι διαφορές. Θα ήθελα λοιπόν τα μέλη να σχολιάσουν και να, υποβάλω και, και να υποβάλλετε και ορισμένες ερωτήσεις και ερωτήσεις. Ο κύριος Κρόιτσμαν έχει το λόγο καταρχήν και νομίζω ότι η κυρία Λεγκρίπ είναι εδώ, σαλτεμόζε, Ρούλε και ίσως και εγώ να λάβω το λόγο στο τέλος. Ε, κύριε Κρόιτσμαν, ε, έχετε το λόγο. Η κυρία Σάλτε Μόζε είχε δείξει το ζήτημα και πάντα ενδιαφέρεται σε θέματα εσωτερικής αγοράς και εποπτείας της αγοράς. Αν εξετάσει κανείς την έκθεση θα δει πρώτον από το 2009 στο 2010 μεγάλη αύξηση, δραματική αύξηση μέχρι 80.000 περιπτώσεις και μετά στη σελίδα 17 84% προέρχονται από την Κίνα αν εξετάσει κανείς ε, ανα εμπόρευμα και αν εξετάσει ανα ε, αποστολή βλέπει ότι είναι 72%. Βλέπει κανείς λοιπόν που βρίσκεται λίγο πολύ το πρόβλημα. Επίσης ενδιαφέρον έχει σελίδα 13 όπου δείχνει υπόθεση πώς, που βρίσκονται οι χώρες μέλη. Η Γερμανία και Μεγάλο, Μεγάλη Βρετανία βρίσκονται πραγματικά ε, στην κορυφή. Αυτό σημαίνει επειδή έχουν καλή εποπτεία της αγοράς ενώ οι υπόλοιπε χώρες κοιμούνται και μια ενισχυμένη συνεργασία. Γι' αυτό έχουμε και ένα πειραματικό, ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να αυξηθεί και η αποτελεσματικότητα των παρεμβασιών μας. Γνωρίζουμε ότι η εποπτεία της αγοράς και επομένως και τα τελωνία είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Και αναλόγως με την δέσμευσή τους, με την παρεμβατικότητά τους, ενδιαφέρον είναι βέβαια και, ενδιαφέρον είναι και η περίπτωση της Ελλάδας, που είναι τελείως εκτός στατιστικής. Δεν κάνω κανένα σχόλιο εδώ, αλλά σας δείχνει που βρίσκονται τα προβλήματα. Ασφαλώς και είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κανονισμό και όχι οδηγία. Βέβαια, <clears throat> Εμείς ζητήσαμε να διεξαχθεί και ακρόαση το Νοέμβριο και το πρόβλημα θα εντοπιστεί περισσότερο στις λεπτομέρειες. Πρέπει να ακούσουμε τους λεγόμενους stakeholder για το πού εντοπίζουν τα προβλήματα, για το δικαίωμα, για παράδειγμα, των ε, ενδιαφερόμενων μερών να ε, τύχουν ακρόασης. Διαβάζοντας τον κανονισμό, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει, εάν έχει αποκαλύψει κάτι ε, το τελωνίο, να καταστραφεί το εμπόρευμα και μετά βέβαια δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει αυτό. Το κόστος της καταστροφής ε, να το αναλάβουν. Το ζήτημα είναι εάν για παράδειγμα στην Κίνα, θα, ε, για περιπτώσεις δηλαδή παραγωγής Κίνας, αν θα λάβει τίποτα από την εταιρεία παραγωγής ως ε, αποζημίωση για, την, για τα έξοδα καταστροφής. Τι γίνεται εάν έχει γίνει λάθος από τα τελωνία ή να έχει γίνει μια παραγγελία μέσω διαδικτύου, παίρνουν τα λεφτά από την πιστοτική κάρτα και μετά δεν λαμβάνει το εμπόρευμα διότι το κατέσχει το τελωνίο. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εμείς θέλουμε να, ε, προστατεύσουμε τον ε, καταναλωτή. Λοιπόν υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις. Τα τελωνία έχει αποδειχθεί από την εμπειρία μπορούν να αποκαλύψουν ε, σχετικά απλές περιπτώσεις ε, παραποίησης. Τι γίνεται με πιο περίπλοκες, για παράδειγμα την τοπογραφία ε, των ηλεκτρονικών chip και ούτω καθεξής. Πώς θα εξασφαλιστεί επίσης ότι για την διαμετακόμιση ε, ορισμένων, για παράδειγμα, φαρμάκων με γενική ονομασία, ότι θα καταλήξουν πραγματικά και στην, ε, στον προορισμό τους. Και οι απλοποιημένες διαδικασίες, όπως είπα και πριν, πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα αυτή, για την καταστροφή τους δηλαδή. Συνοψίζοντας, θέλω να πω ότι θα εξετάσουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, θα τις συζητήσουμε είναι βέβαια απαραίτητο αυτό, βλέπουμε και ε, τις αυξήσεις των αριθμών, το γεγονός δηλαδή ότι η Κομισιόν προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού της. Στην ακρόαση ας συζητήσουμε τις λεπτομέρειες, γιατί εκεί θα σημειώνονται τα περισσότερα προβλήματα. Βέβαια, προς το συμφέρον του καταναλωτού, αλλά και προς το συμφέρον του δικαιούχου της διανοητικής ιδιοκτησίας αν εξετάσει κανείς πού σημειώνονται οι παραβιάσεις, υπάρχει μια στατιστική και βλέπει κανείς ότι είναι πολύ συχνά τα τσιγάρα, το ίδιο όμως τα παιχνίδια, ε, εμπορεύματα, ενδυμασίες, ενδύματα, επίσης ακριβές τσάντες χειρός κλπ. Ότι γίνεται κάτι είναι καλό, θα τα συζητήσουμε όπως είπα και ελπίζουμε. Είναι χαρακτηριστικό, είναι, είναι, είναι κύριο θέμα προστασίας του καταναλωτού. Αλλά βέβαια όχι μόνο προστασία του καταναλωτού, προστασία και των επιχειρήσεων που έχουν το ενδιαφέρον, έχουν το συμφέρον, ε, τα υψηλής ποιότητας εμπορεύματά τους, τα οποία προκύπτουν μετά από πολλή επένδυση και σε έρευνα και ανάπτυξη κλπ. Εν τέλει την πληρώνει ο καταναλωτής συχνά. Αλλά όχι μόνο. Όταν κάποιος έρχεται από τις διακοπές ε, στην Αλοδαπή και ε, είναι υπερήφανος για μια ωραία τσάντα που αγόρασε, καμιά φορά δεν γνωρίζει καν ότι help if we don't have the sufficient resources uh, in the customs to take uh, care of the new regulation. Uh, Do we have, do the member states have uh, sufficient resources to take care of this uh, area? Because if they don't, then new legislation will. Τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να επομιστούν όλα αυτά που θα τους δείσει η νέα νομοθεσία. Αλλιώς τι να την κάνουμε τη νέα νομοθεσία και το νέο κανονισμό. Πρέπει να τον επιβάλλουμε και χρειάζονται για να τον εφαρμόσουμε πόροι επιπλέον. Τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας, τα κράτη-μέλη τα γνωρίζουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλε, έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε. Έχω και εγώ μερικέ ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, στα αγγλικά τώρα κυρία Ρούλε, αναφέρατε τρία προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι ο κανονισμό δεν καλύπτει κάποιες παραβιάσεις ε, των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία. Ποιοι είναι αυτοί οι τομεί δηλαδή που δεν καλύπτονται. Δεύτερον, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Σάλτεμος, αν διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή και δεν φροντίσουμε να έχει μεγαλύτερη στελέχωση η αρμόδια υπηρεσία, δεν θα έχει νόημα. Κοίταξα και τις στατιστικές σας και καμιά φορά αναφέρεται κάποια λοιπά εμπορεύματα. Τι, τα λοιπά αυτά τι είναι, ποια είναι τα λοιπά προϊόντα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αξία τους πολλές φορές. Τα λοιπά αυτά ποια είναι. Και μια τρίτη ερώτηση. Το παράλληλο εμπόριο που δεν καλύπτεται ακόμα από τον κανονισμό θα το συμπεριλάβετε εκεί. Είναι μεγάλα τα ποσά και αφορούν ε, και φάρμακα. Έτσι δεν είναι. Και έχω ένα ερωτηματικό. Γιατί πρέπει ξαφνικά να καλύπτεται από εδώ και μπρο και δεν καλυπτόταν μέχρι σήμερα. Ελπίζω να μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση και γι' αυτό. Αυτά. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω μερικά στα όσα είπαν οι συνάδελφοί μου, αν μου επιτρέπετε. Ένας από τους τομείς που θα μας ενδιαφέρει για να καταλάβουμε τι γίνεται, να μάθουμε, ε, είναι αυτό το τελευταίο που είπε η κυρία Ρούλε. Θα μπορούσαμε να σε εξηγήσετε και πάλι τους νέους τομείς που επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Γιατί είναι λίγο πιο δύσκολο να το καταλάβουμε σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό. Και τώρα είναι σημαντικό στοιχείο της πρότασης, όπως είπατε και εσείς στη μελέτη αντικτύπου. Ένας από τους λόγους αλλαγής είναι ότι τα θέματα διανοητικής διακρισίας και δικαιωμάτων έχουν εξελιχθεί και έχουν μπει και νέα στοιχεία, για παράδειγμα γεωγραφικές ενδείξεις. Και ίσως θα ήταν χρήσιμο να μας δώσετε κάποιο χάρτη διασταυρωμένες ε, ε, ενδείξεις και στοιχεία για να ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Στη συνέχεια θα με ενδιαφέρει να μάθω γιατί είχαμε και σχετική εμπειρία στην Επιτροπή μας από επισκέψεις που κάναμε στο Ρότερνταμ και στην Αμβέρσα δεν πήγαμε μάλιστα και στη Σανκάη και αλλού. Και είδαμε και εμπορεύματα παραποιημένα που είχαν κατασχέσει στη Σανγκάη. Οι τελωνιακές αρχές. Και αν δεν απατώμε, να μην κάνω και λάθος στην ορολογία, η εκτίμηση κινδύνου είναι αυτή που μας ενδιαφέρει. Η πρώτερη γνώση και πληροφόρηση για να ξέρουμε ε, ποια είναι τα ύποπτα φορτία και αποστολές. Έτσι το λέτε, σε εκτίμηση κινδύνου. Αυτά τα στοιχεία θα βοηθήσουν ε, τις αρχές ε, για να κάνουν τους ελέγχους και να αναλάβουν τη δράση. Α, πήγαμε και στην Ινδία, ξέχασα να πω. Δηλαδή γυρνάμε αρκετά και κυκλοφορούμε και κοιτάζουμε. Οι τελωνικέ αρχές μας αναφέρουν αυτά τα στοιχεία ε, του κινδυνού, της εκτίμησης κινδυνού της πρώτερης πληροφόρηση, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των φορτίων και των εμπορηματοκιβωτίων που μπαίνουν σε ένα λιμάνι και πρέπει να ξέρεις ποιο θα πας να ελέγξεις. Σε αυτό το νέο κανονισμό υπάρχουν κάποια στοιχεία που να βοηθήσουν τις αρχές για να δρουν εκ των προτέρων, ε, να ζητούν από τους μεταφορείς ε, και του, ε, πληροφορίες για να μπορούν να δρουν σωστά. Και μετά τι γίνεται μετά την κατάσχεση. Έχουμε την αίσθηση ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες σημάτων και δικαιωμάτων ε, δείχνουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα όσο και αιμονή στην αντιμετώπιση αυτών των ε, καταστάσεων, έχουν πιο αξιόπιστες πηγές, πιο γρήγορες πηγές και σε ό,τι αφορά την κατάσχεση και την καταστροφή των εμπορευμάτων. Και επίσης δεν κατάλαβα από τόσα μας είπατε εάν ε, θα προτείνεται νέα μέτρα για την ανταλλαγή πληροφοριών, για τη διαβίβαση πληροφοριών και τη ταχύτητά της. Γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο ε, κάποιος ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί εγκαίρως και αν πρέπει να αναλάβει την αποστολή της καταστροφής μιας παρτίδας. Γιατί ψάχνουν να βρουν ποιος θα τους ε, δώσει την άδεια να καταστρέψουν ένα φορτίο, δεν θέλουν να το καταστρέψουν. Αυτά. και ήταν δύσκολο πολλές φορές στην παρουσίασή σας να αντιστοιχίσουμε το νομοθετικό πλαίσιο που μας προτείνεται με τις αγωνίες και τις ανησυχίες των ενδιαφερομένων επιτόπου. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλει κανένα άλλο το λόγο. Καλώ. Τώρα δεν ξέρω ποιο θέλει να απαντήσει πρώτο. Εσείς, μάλιστα. Very um, ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα σημαντικά ερωτήματα τα οποία υποβάλλατε. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει τη συλλογιστική μας γιατί προσπαθούμε να στοχοθετήσουμε σωστά τα προβλήματα. Για να απαντήσω στον κύριο Κρόιτσμαν θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να γίνουν ενδελεχείς συζητήσεις για την ουσία της πρότασης και ελπίζω να, σας, να μπορέσουμε να σας την παρουσιάσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για να δείτε πού ε, έγκυνται οι ανησυχίες μας. Και επίσης μπορούμε να σας δώσουμε και οποιασδήποτε πληροφορίες επιθυμείτε. Τώρα σε σχέση με το θέμα της προστασίας των καταναλωτών έναντι των συμφερόντων των βιομηχανιών και επιχειρήσεων, νομίζω από, από ό,τι κατάλαβα από το σχόλιο, τα σχόλια της κυρία Σάλτε Μόζε, πρωτίστως μας ενδιαφέρει η προστασία του καταναλωτή. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αγοράσει αγαθά από το διαδίκτυο. Αλλά παράλληλα δεν πρέπει να διακυβεύεται η ασφάλεια του διότι πολλές φορές εξαπατώνται οι καταναλωτές από την αγορά μέσω διαδικτύου. Βεβαίως, το άλλο στοιχείο είναι τα ε, συμφέροντα των επιχειρήσεων και αυτό που μας ενδιαφέρει μέσα στα πλαίσια της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι να προωθήσουμε την παραγωγικότητα, άρα προωθούμε και το συμφέρον των επιχειρήσεων και των εμπόρων και του εμπορικού δικτύου που έχει ειδικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Σαλτεμόζ ρώτησε κατά πόσο τα κράτη-μέλη γνωρίζουν ότι υπάρχει σωρία προϊόντων τα οποία ε, φτάνουν στις ε, τελωνιακές αρχές. Οι τελωνιακές αρχές κοινοποιούν τα δεδομένα και ε, οι τελειωνιακές ε, αρχές ήταν αυτές που μας μίλησαν για τις ταχυδρομικές αποστολές αυτών των αγαθών και όπως ξέρετε στη, στα ταχυδρομεία δεν υπάρχουν ε, τελωνιακές αρχές, γι' αυτό πρόκειται για μία ε, ιδιαίτερα φορτωμένη διαδικασία. Κατανοούμε την κατάσταση και ελπίζω το Συμβούλιο θα συμφωνήσει ότι θα πρέπει να απλουστεύσουμε τη ζωή των τελωνιακών αρχών. Μιλήσατε για τους ε, πόρους που υπάρχουν στα τελωνία. Αυτό δεν αφορά άμεσα την Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο σχόλιο. Σήμερα δεν μπορούμε να ανοίξουμε όλα τα κουτιά ε, όλες τις αποστολές που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ανάλυση, γι αυτό, ε, που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δεν μπορούμε να προβούμε σε μια ενδελεχή ανάλυση κινδύνου. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κίνδυνο μέσα στα πλαίσια της TAXUD. Στη νομοθετική πρόταση υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία έχουμε εισαγάγει έτσι ώστε τα τελωνία να κατέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες. Βλέπετε στο κεφάλαιο της εφαρμογής και της συμπλήρωση της αίτηση, εδώ γίνεται μία διασάφιση των πληροφοριών που θα πρέπει να δοθούν προς τα τελωνία και εδώ θα πρέπει να υπάρχει πλήρης